Εμεί υπερψηφίσαμε με πλειοψηφία. Εκεί γίνεται μια πρόβλεψη για τις διαπραγματεύσεις, τις τριμερείς διαπραγματεύσεις σε σχέση με μέτρα στήριξης του γεωργικού τομέα ε, σε σχέση με την, ε, με την επιβολή δασμών. Ε, δεν θα πρέπει ο τομέας αυτός ε, να πληγεί από τον ε, πόλεμο το οποίο θα ξεκινήσει η το Ενωμένο Βασίλειο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κυρία Γκλέρα. Η κυρία Ζανό. Thank you, Chair. I voted in favor of... Uh, εγώ υπεψήφισα την πρόταση αυτή γιατί υποστηρίζει τα προγράμματα για τους νέους. Αλλά για το 2015 είμαι κατά. Αυτοί που συμφωνούν να δίδονται ε, που το υπεψήφισαν δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες για το πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά γιατί πρόκειται για προϊόντα τα οποία είναι πραγματικά απαράδεκτα, είναι προγράμματα και ισχυρισμοί ε, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να στηριχθούν. Και κανένας δεν μπορεί φυσικά να γνωρίζει κανείς τις υπερβολές, στη Λετωνία σαν παράδειγμα, είναι σαφές ότι κυκλοφορούν στοιχεία και πληροφορίες που προέρχονται από την ίδια πηγή ε, τα οποία αφορούν τη Λευκορωσία αλλά δυστυχώς ε, τα στοιχεία τα οποία έχει δώσει η χώρα μου δεν έχουν ε, εκπροσωπηθεί ή τουλάχιστον δεν έχουν παρουσιαστεί με τον σωστό τρόπο. Ευχαριστώ ο κύριος Πάλμερ, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Και εγώ θέλω να αναδείξω την ε, στήριξη του Erasmus Plus. Θα ήθελα όμως πάλι να μιλήσω για την αμφιβολία και την ανασφάλεια λόγω του Brexit ε, το οποίο όμως συνεμετέχει στο Εράσμους. Οφελήθηκαν χιλιάδες Βρετανοί νέοι και φέτος και τα προηγούμενα χρόνια από το Εράσμους. Η Ένωση των Πανεπιστημίων είδα, διαπίστωσε ότι 94% των πανεπιστημίων δεν θα μπορούσαν να ε, συμμετέχουν στο Εράσμος αν δεν ε, υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να συνεχίσουμε στο Εράσμος και μετά το 2020. Ε, καλώ τη Βρετανική κυβέρνηση να διευκρινίσουν ότι θα συμμετέχουν και στο μέλλον στο Εράσμους και να ρωτήσουν τους νέους ε, αν ε, επιθυμούν ε, αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ. Όπως και ο συνάδελφος ε, Κάρθη μιλάω στην μητρική μου γλώσσα. με χαρά υποστήριξα αυτές τις προτάσεις γιατί είναι αξιόλογες. όταν ε, τιμήσεις τους νέους ε, θα, σε προσεγγίσουν. Ε, είναι καλό το Erasmus Plus, είναι δυνατότητα για κινητικότητα. Επίσης, οι συστάσεις για την κλιματική αλλαγή και η σχετική πάλι είναι αξιόλογες. Πρέπει να, το κάνουμε, να τα κάνουμε αυτά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Είναι ζωτική σημασία να δώσουμε σε όσους πλήττονται, τις χώρες που περισσότερο πλήττονται, να δώσουμε στήριξη. Ε, με χαρά λοιπόν στήριξα τις προτάσεις αυτές γιατί θα βοηθήσουν την Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελείωσαν οι επεξηγήσεις για την έκθεση Χολμάιερ και Ρουμπιάλ. Τώρα, έκθεση Σάρβαμα, απαλλαγή 2017, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξη για το Άσυλο. Ο συνάδελφος Ρος κάνει την αρχή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το... Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία πρέπει να διασφαλίζει ότι η πολιτική ασύλου ε, στα κράτη-μέλη θα ε, συμμορφούνται προς τους ε, κανόνες. Λειτουργήσε όμως ε, με διοντολογικά ε, άσχημο τρόπο. Μετά το 2016 και το 2017 η Όλαφ ανακάλυψε ότι ε, οι διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων ήταν λάθος, υπήρχαν κακοδιοίκηση, και άλλες ατασταλίες, προβλήματα με την πολιτική προσλήψεων, ε, παρενόχληση, εκφοβισμός ε, στο προσωπικό. Ε, δεν μπορούμε να εγκρίνουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς θέλουμε απόλυτη διαφάνεια εδώ και γι' αυτό δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε στην απαλλαγή. Ο συνάδελφος Πόλτσακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σίγουρα η υπηρεσία για το άσυλο είναι μια προτεραιότητα στον τομέα της ασφάλειας ε, ενάντια στα κύματα βίας από πλευράς κάποιων προσφύγων στην Μόλτα, Μάλτα για παράδειγμα. Ε, αυτό είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο όμως είναι αυτό που συνέβαινε στην υπηρεσία εγώ υποστήριξα την, ε, το ψήφισμα για την απαλλαγή για το 17, αλλά αυτή η περίοδος σχετίστηκε με πολλά προβλήματα στις δημόσιες συμβάσεις και άλλα προβλήματα. 7,7 εκατομμύρια ευρώ, 10% δηλαδή των πληρωμών της υπηρεσίας ήταν λανθασμένες Επίσης υπήρχαν προβλήματα με τις ε, προσλήψεις. Ο εκτελεστικός διευθυντής πέρσι παρατήθηκε. Εύχομαι στη νέα διεύθυνση κάθε επιτυχία ώστε να γίνει μια, αυτή η απαραίτητη για μας υπηρεσία διαφανής. Ευχαριστώ και ο συνάδελφος Κέλλη. Εγώ, όπως και ο κύριος Πόλτσακ, ε, ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής Ακόμα και το ελεγκτικό συνέδριο μας συνέστησε να εγκρίνουμε γενικά. Υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις σε πληρωμές, υπήρξαν επίσης και κάποιες ε, καταχρήσεις στον τομέα ε, των κοινοτικών κονδυλίων. Υπήρξαν επίσης και ε, απαράδεκτες μορφές bullying εις βάρος του προσωπικού και γι' αυτό ακριβώς όπως και ο κύριος Ρούς θα πω ότι απαιτείται πλήρης διαφάνεια και θα πρέπει να το απαιτήσουμε στο μέλλον αυτό. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κέλλη. Ολοκληρώνεται εδώ η διαδικασία επεξηγήσεων ψήφου για την έκθεση αυτής και ακολουθούν επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση της κυρίας ε, Μουνιώθ για την απαλλαγή προς το Συμβούλιο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ που μου δάσατε το λόγο, Πρόεδρε. Σχετικά με την απαλλαγή του Συμβουλίου Υπουργών και του Συμβουλίου γενικότερα. Εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις αρμοδιότητες που έχουμε, τις εξουσίες που έχουμε στον τομέα του προϋπολογισμού και στον τομέα του ελέγχου του προϋπολογισμού και βλέπουμε ότι είναι απτή μια διοργανική θα έλεγα ένταση ανάμεσα στο Συμβούλιο ε, και το Κοινοβούλιο. Δεν θα πρέπει να αμφισβητείται όμως ε, η δυνατότητα την οποία έχουμε. Αν θέλουμε πράγματι ο προϋπολογισμός να είναι διαφανής και να ελέγχεται, είναι σαφές ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε το ρόλο μας και να μην υπάρχουν στρεβλώσεις στην κατανομή των εξουσιών. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πόλτσακ. Ακολουθεί ο συνάδελφος κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω την πρόταση άρνησης χορήγησης απαλλαγής του Συμβουλίου Υπουργών. Ε, το Συμβούλιο είναι ένα απέσιο σώμα, είναι μυστικοπαθές και βλάπτει την εμπιστοσύνη του κοινού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ντρέπονται για την κατάσταση αυτή. Αλλά η άρνηση της απαλλαγής ε, είναι λάθος, γιατί τότε θα αρχίσουν να επιτίθενται στο δικό μας προϋπολογισμό και θα μπούμε σε ένα άχρηστο πόλεμο που θα χάνουν όλοι το χρόνο τους. Ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση της μυστικοπάθειας αυτής είναι να υπογραμμίζουμε συγκεκριμένα παραδείγματα σπατάλης με εξωτικές συναντήσεις των Υπουργών όπου δεν έχουν και πολλά να συζητήσουμε. Λοιπόν, αυτός θα ήταν ο σωστός τρόπος να τους δείξουμε με το δάκτυλο και να τους ζητήσουμε να χρησιμοποιούν τα χρήματα των φορολογουμένων με ορθό πλέον τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Νιούτον Ντάν. Τελευταίος ομιλητής από τον Σον Κέλλη. Είναι σαφές ότι το Συμβούλιο δεν έδωσε τις απαντήσεις, τις γραπτές ερωτήσεις που είχαμε καταθέσει σαν Κοινοβούλιο και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου δεν ήταν καν παρόν στην ακρόαση την οποία οργανώσαμε. Γι' αυτό λοιπόν οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαρτίου 2019 δεν έγιναν αποδεκτές. Αυτό είναι απαράδεκτο και γι' αυτό θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στο Συμβούλιο ότι θα πρέπει τις θέσεις μας να τις λάβει σοβαρά υπόψη. Όλα τα όργανα της Ένωσης πρέπει να είναι διαφανή, πρέπει να είναι υπόλογα στους πολίτες της Ένωσης γιατί τους εμπιστεύεται το κοινό και τους χρηματοδοτεί και θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους πλέον. Και είμαι ικανοποιημένος που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει στο θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η διαδικασία επεξηγήσεων ψήφου. Και φτάσαμε και στο τέλος της ημερήσιας διάταξης. Ε, εύχομαι σε όλους που παρευρίσκονται ακόμα εδώ. Καλή όρεξη μέχρι τις 3 το απόγευμα.